Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίσω την έναρξη συνεδρίασης ε, της Επιτροπής Ελέγχου Προπλογισμού για σήμερα. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι χθες όπως και χθες μάλλον είναι δημόσια συνεδρίαση με τις αντίστοιχε γλώσσες και μάλιστα μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Αρχίζουν ψηφοφορίες λοιπόν. which is today? Which one? Und zwar sind äh, heute auf der Agenda die Entlastung. Έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη την απαλλαγή των οργανισμών με εισηγητή τον κύριο Γερμπραντή. Χερμπράντη. Επιθυμείτε να λάβει το λόγο κύριε εισηγητά. Έχετε ακόμα κάποια τροποποίηση να επισημάνετε. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, γιατί είναι βέβαια και αρκετά μακρά η ψηφοφορία που έχουμε μπροστά μας. Ωστόσο, να κάνω λίγα σχόλια. Πρώτα, να ευχαριστήσω όχι μόνο τους ίδιους τους οργανισμούς για τη συνεργασία τους. Μέχρι ακόμη εχθές το βράδυ ήμουν σε επαφή με ορισμένους οργανισμούς για να ρυθμίσουμε ας πούμε, τα τελευταία εκκρεμή θέματα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές που έδειξαν πνεύμα συνεργασίας και τέλος, το προσωπικό της ε, γραμματείας της Επιτροπής που πραγματικά σκοτώθηκε στη δουλειά για να φτιάξει όλες αυτές τις εκθέσεις που θα ψηφιστούν σήμερα. Τους ευχαριστώ λοιπόν πραγματικά για τη σκληρή δουλειά, μάλιστα και στις διακοπές των Χριστουγέννων. Έχω τώρα ορισμένα σχόλια για τη σημερινή ψηφοφορία Πολλή δουλειά έγινε και παρασκηνιακά, σε συνεργασία και με τους οργανισμούς και η πίεση της αναβολής της απαλλαγής καμιά φορά παίζει όντως σημαντικό ρόλο για να οθήσει τους οργανισμούς να εκτελέσουν το έργο τους. Πάντως είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά που έγινε και γι' αυτό η πρότασή μου είναι να χορηγηθεί απαλλαγή σε όλους τους οργανισμούς και σε όλα τα joint undertaking. Παρ' όλα αυτά, ορισμένα σχόλια έχω για ορισμένους από αυτούς. Αρχίζω με τις ε, joint undertakings, τις κοινοπραξίες. Είναι η ε, είχαμε εκεί έκθεση από το ελεγκτικό συνέδριο για τη στρατηγική μετά τον έλεγχο. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένες διαφθορτικές αδυναμίες στο σύστημα ελέγχων τους και λόγω του τρόπου χρηματοδότησής τους. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έλαβα επιβεβαίωση από την Επίτροπο Κρούς που είναι ευθύνη στις αυτές, αυτές οι κοινέ επιχειρήσεις για ότι θα αντιμετωπίσει αυτές τις διαρθρωτικές αδυναμίες. Και για το λόγο αυτό, λόγω της διαβεβαίωσης αυτής, προτείνω απαλλαγή. Για τους οργανισμούς τώρα θα αναφερθώ μόνο σε τρεις. Πρώτο για την ασφάλεια των εναέριων μεταφορών. Όπως συζητήσαμε και εδώ στην Επιτροπή, είχα ανησυχίες σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, όχι εντός του οργανισμού, αλλά μεταξύ του Διοικητικού της Συμβουλίου και του οργανισμού. σε εκτεταμένες επαφές και με τον εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού και με τον πρόεδρο του Management Board και χθε έλαβα την διαβεβαίωση από την επικεφαλής του Managing Board ότι έλαβαν κοινοποίησει για τις συγκρούσεις συμφερόντων και έχουν λάβει τώρα τις περισσότερες από τις ε, υπογεγραμμένες δηλώσεις συμφερόντων των μελών του Συμβουλίου και φαίνεται ότι οφείλεται μοναχά σε τυπικούς λόγους, σε γραφειοκρατικούς λόγους ότι δεν έχουν λάβει όλες τις ε, δηλώσεις και ότι δεν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόβλημα. Γι' αυτό και προτείνω και εδώ απαλλαγή. εν τέλει, ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα αλλά και ο Οργανισμός για το Περιβάλλον, ως γνωρίζουμε, και, οι δύο, και για τους δύο μάλλον εκκρεμούν έρευνες του Όλαφ. Άλλωστε και για μας ε, και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι έχουμε έξι εκκρεμείς υποθέσεις το ίδιο το Κοινοβούλιο. Εν γέννη πάντως, οφείλω να πω ότι έρευνα του Όλαφ καθεαυτήν δεν αποτελεί λόγο ε, άρνησης της απαλλαγής. Είναι ξεχωριστές ε, ιστορίες αυτές και ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα προς πληροφόρησή σα λέω ότι ο Όλαφ έκλεισε την έρευνα χωρίς να κάνει καμία σύσταση, αλλά αυτό είναι καλό νέο για τον οργανισμό. Για τον οργανισμό περιβάλλοντος ενημερωθήκαμε από τον διευθυντή του Όλαφ την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της έρευνάς τους όχι για το περιεχόμενο, αλλά ο εκτελεστικός διευθυντής με πληροφόρησε για το περιεχόμενο της έρευνας. Κανένα από τα θέματα της τρέχουσας αυτής έρευνας δεν αναφέρεται στο έτος 2011. Και εδώ βέβαια μιλούμε για απαλλαγή για το 2011, ώστε στην έρευνα του Όλαφ δεν αναφέρεται τίποτε στο έτος αυτό. Ούτε το ελεγκτικό συνέδριο, ούτε ο εσωτερικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν βρει οτιδήποτε που να μην ευθυγραμμίζεται με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Και γι' αυτό συνιστώ στην παρούσα Επιτροπή να υπερψηφίσει τη χορήγηση της απαλλαγής του Οργανισμού Περιβάλλοντος και να μην την αναβάλει μέχρι φέτος το φθινόπωρο. Αυτά είναι τα σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και βεβαίως όπως είπα η ψηφοφορία θα είναι μακρά. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά, λέει ο για τα συμπληρωματικά αυτά σχόλια. Τα μέλη της Επιτροπής είχαν επαρκή χρόνο για να εγκύψουν στο θέμα, ώστε να μπορούν να ψηφίσουν όπως το υπαγορεύει η συνείδησή τους. Αρχίζουμε τώρα την συζήτηση. Πρώτο, το υπαριθμό 39. απαλλαγή του Άρτεμις. Είναι στο υπαριθμό 8. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες. Αρχίζω. Πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία θα χρειαστεί να κάνουμε και ονομαστικές ψηφοφορίες ηλεκτρονικές δηλαδή. Θα κάνουμε πρώτα ένα τεστ της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αρχίζει τώρα. Αρχίζει. Σας ευχαριστώ, ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρας. Ωραία λοιπόν. Βλέπετε το αποτέλεσμα. 23 ψηφίζουν λοιπόν. Έχουμε τώρα τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, Α κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 8. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπαριθμούν 10 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε τροπολογία 10 πρόκειται για το item 8 τελειώσατε, ε, ψηφίσατε όλοι παρακαλώ τέλος, εγκρίθηκε λοιπόν σαφώς τώρα τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 13 13 ως προσθήκη Μόνο όμως εφόσον εγκριθεί η 12, αλλά η 12 απορρίφθηκε. Α, το ψηφίζουμε λοιπόν. Καλά, ψηφίζουμε την 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται υπαριθμών 14 υπέρ κατά α εκπίπτει αυτή ναι ναι η 12 έχει η 12 έχει εγκριθεί αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό καλά η 14 εκπίπτει εν πάση περιπτώσει τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εφόσον εγκρίνεται εκπίπτει 28 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές. Παρακαλώ επαλήθευση. Τροπολογία 30. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, επαλήθευση. 32. Επαλήθευση ηλεκτρονική. 32. Ψηφίσατε παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συνεχίζω, η 34 εκπίπτει, τροπολογία 35 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση παρακαλώ, 35 επαλήθευση. Ψηφίσατε. Τέλος της ψήφου. εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Εκπίπτει. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 41 υπέρ κα, κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ 41 ψηφίσατε πέρασε Α, βλέπω ότι το Λαϊκό Κόμμα έχει μία ψήφο παραπάνω από όσους δικαιούται. Ποιος θα αφαιρέσει. Ωραία λοιπόν. Πέρα στη ψήφο. Εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ επαλήθευση. 45. Ψηφίσατε. Τέλος. εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται αλλά προτιμώ να γίνει ονομαστική ψηφοφορία γιατί δεν συμμετέχετε όλοι. 47 ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ ωστόσο όλοι να συμμετέχετε στην ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεν ήταν ωστόσο βέβαια και τόσο ε, εύκολο να το διακρίνει κανείς 13 υπέρ 12 κατά. Κύριε Γκάιερ. Έχουμε τον κύριο Ιβαν εδώ, ο οποίος ε, έχει ξεχάσει την κάρτα του, ή δεν την έχει μαζί του, και θα ψήφιζε κατά. Α, λυπάμαι πολύ να μάθετε να χάνετε. δεν παρενέβη μέχρι τώρα, αλλά τώρα είναι κρίσιμο και γι' αυτό παρεμβαίνω. Τότε θα ξαναψηφίσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Θα έρθει η ηλεκτρονική σας κάρτα, μάλιστα. Είναι καθοδόν. Επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω την ψηφοφορία. Τροπολογία λοιπόν 47. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ε, ψηφίσατε όλοι, παρακαλώ. Τέλος. Ορίστε λοιπόν το αποτέλεσμα. Λυπούμε πολύ. Χαίρομαι που ξυπνήσαν όλοι, λέει ο κ. Γκάιερ, τουλάχιστον. Τροπολογία 48. ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση. 53. Ψηφίσατε παρακαλώ. Όχι ακόμη. Τέλος. Ο κύριος Ιβαντή ψηφίζει. Έχετε την κάρτα σας τώρα. Ναι ή όχι. Υπέρ ή κατά. Είστε κατά. Άρα ισοψηφία 13 προς 13. Απορρίπτεται. 54. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αυτή. Τροπολογία 55 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 υπέρ, Α, θέλετε επαλήθευση 58. Ωραία. Επαλήθευση 58. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Κύριε Ιβάν, Κατά. Άρα λοιπόν η ισοψηφία 13 προς 13 απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει. Ψήφισατε όλες και όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά άποχες δεν είναι σαφές 62 επαλήθευση παρακαλώ 62 ψηφίσατε όλοι πέρασε εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 είναι γλωσσικής φύσεως, δεν ψηφίζεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. 74 ηλεκτρονική επαλήθευση. Τέλος της ψήφου. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 έως 79 εκπίπτουν. Σωστό είναι αυτό. Έχει καλώς. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει. Τροπολογία 81. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας. Α, συγγνώμη. Σαφώς εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. 84. Επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίσατε. Πέρασε. Έχει καλός λοιπόν. Άρα παρακαλώ όλοι να ψηφίζετε τάσω της χειρός. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται αυτή 89 υπέρ <clears throat> κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτή 90 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται ο 91 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται και αυτή. 94 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Αυτό δεν είναι σαφέ. 94 ηλεκτρονική παρήθεση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Απέριφθη. Ακολουθεί η 95. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 98 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται με κάποιο δισταγμό λέει ο πρόεδρος αλλά ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά αρχίζει η ψήφος τέλος εγκρίθηκε όντως τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται απασχόλησης ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απασχόλησης δύο υπέρ με η κυρία Σέντερ χωρίς μικρόφωνο έμπλ, έμπλ είναι στα αγγλικά έμπλ δύο. είμαι στις έμπλ τροπολογίες δηλαδή Επιτροπής Απασχόλησης. Υπάρχουν δύο τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Οι δύο της Επιτροπής Απασχόλησης. Τέλος. Εγκρίνεται. Το Apple 3, αλλά είναι out of scope, είναι εκτός ε, πεδίου εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Αλλά χρειάζεται μάλλον να ψηφιστεί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εμπολ 4, αλλά δεν προβλέπεται ψηφοφορία εδώ. Για την 5 ισχύει το ίδιο. Ψηφίζουμε λοιπόν την επιστοπή τη Περιβάλλοντος, την υπαρχόν 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. Συνεχίζω στην NV6, περιβάλλοντος 6, Περιβάλλοντο 6 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπάρχει μια αλλαγή τώρα στην επιτροπή που έχει υποβάλει, είναι η θεμελιωδών ελευθεριών. Λίμπε ένα λέει ο πρόεδρος. Έχει βάλει μείον. Ο εισηγητής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζω. Λίμπε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και λίμπε 4 υπέρ κατά αποχές αν εγκρίνεται και αυτή. Θα ψηφίσουμε τώρα το ψήφισμα. Πριν το ψήφισμα... Α, η κυρία Σέντερ. Την τροπολογία 80, γιατί είμαι λίγο βραδίστροφη σήμερα το πρωί. Η τροπολογία 80 ζητούσε απάλληψη, την υπερψηφίσαμε όμως. Και μετά ήταν η 81 που ετέθη προς ψήφιση και την εγκρίναμε. Ε, δεν γίνεται όμως. Γιατί υπάρχει και η παράγραφος 32. Ε, ναι, το έγραφε ο κατάλογος φοφορίας μου λέει ο πρόεδρος, όχι ο δικός μου λέει η κυρία Γιάλα. Εγκρίναμε την 80 και 81 καταπίπτει. Ναι, δεν το έγραφε ο κατάλογος, έπρεπε να το διορθώσουμε, έχετε δίκιο. Τώρα όμως... Ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία επί της απαλλαγής του θέματος του 8. Item 8. 8. Ηλεκτρονικά, ονομαστική ψηφοφορία δηλαδή. Αρχίζει, ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. η ομάδα ECR των Βρετανών Συντηρητικών έχει μία ψήφο παραπάνω από τη δικαιούται. Πέρας. Εγκρίνεται. Okay, we continue with item 8. Nine, sorry. We just finished eight and we continue with nine. Συνεχίζουμε λοιπόν με το 9. Μόλις τελειώσαμε το 8, συνεχίζουμε με το 9. Συμφωνείτε? Κάτι δεν λειτουργεί? One dropped out, colleague A. Pink. But now it seems that they are only three. Strange. Uh-huh. Yeah, sorry. Mr. President, uh, perhaps... Κύριε Πρόεδρε, Ίσως δεν γνωρίζετε, η κυρία Αντρέα Σένα την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε στην ομάδα μας, ε, εντάχθηκε στην ομάδα μας ε, και επομένως έχουμε τρεις ψήφους πλέον. Ε, ενδεχομένως να κάποια από αυτές τις τρεις να είναι και αποφασιστική ψήφος. Ίσως δεν έχει... Εντάξει, λοιπόν, να επαναλάβουμε την τελική ψηφοφορία επί του σημείου 8. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν η οποία άρχεται τώρα. Everybody voted. Εψήφισαν όλοι. Δεν λειτουργεί. I was too quick. Vote closed. Τα είπα πολύ γρήγορα μάλλον λέει ο Πρόεδρος. Εντάξει. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με το 9, παράγραφος 1. Ταυτόσιμες τροπολογίες 1 και 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Εγκρίνεται μάλλον. Η τρία καταπίπτει. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επ' αυτού του σημείου. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται σαφώς. Περνάμε τώρα. We need a final vote now. Yes. On everybody. Motion of a resolution now. On which one? of Yeah. Okay. There are no amendments. Δεν υπάρχουν τροπολογίες, ε, αλλά πρέπει να κάνουμε την ε, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο των λογαριασμών. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, λοιπόν. Electronic vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. This one? Just this If we grant this charge, this is automatic. Okay. That falls. Okay. But we still do the final vote, and we did. And what is this? now we go to motion for a resolution. Yep. Okay. We continue with the motion for a resolution. And, uh... Λοιπόν, έχουμε το ψήφισμα και ψηφίζουμε τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε λοιπόν με το σημείο 10. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Ε, λοιπόν, αυτό εγκρίθηκε και τώρα έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο των λογαριασμών. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψήφισμα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημείο 11. Τροπολογία 1 και τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Επί της απόφασης. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της απόφασης άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο των λογαριασμών άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν, άρχεται τώρα. Ψήφισαν όλοι, τέλος. Um, we go back to εάν επί του σημείου 10, εάν η, ο κατάλογος ψηφοφορίας μου είναι σωστός, ε, έπρεπε να υπάρχει μία τροπολογία. Κάναμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία, ε, αλλά δεν ψηφίσαμε αυτή την τροπολογία. Ναι, εγκρίναμε, την εγκρίναμε την τροπολογία αυτή. Ε, λοιπόν, ψηφίζοντας υπέρ της απαλλαγής, η τροπολογία για μετάθεση καταπίπτει και επομένως από τη στιγμή που η πλειοψηφία υπερψήφισε την ε, απαλλαγή ε, τότε δεν υπήρχε λόγος να ψηφιστεί η τροπολογία και επομένως προχωρήσαμε άμεσα στην ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο των λογαριασμών και για το ίδιο το ψήφισμα. Σημείο 12. Η τροπολογία 3 καταπίπτει. Ψηφίσαμε ήδη ηλεκτρονικά για την απαλλαγή, επομένως τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε επί της προτάσεως κλεισίματος των λογαριασμών. Εκεί έχουμε την τροπολογία 4 και την τροπολογία 5. Ο εισηγητής θέλει να πει κάτι. Δεν ψηφίσαμε για το 12 ακόμα. Ψηφίσαμε όμως για τις τροπολογίες 1 και 2 οι οποίες εγκρίθηκαν. Επομένως, ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αποφάσεως ε, περί απαλλαγής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την πρόταση για κλείσιμο των λογαριασμών. Τροπολογίες 4 και 5. Α, όχι, αυτές καταπίπτουν. Επομένως, έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία απευθείας για το κλείσιμο των λογαριασμών. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ωραία. Για το ψήφισμα υπάρχουν τροπολογίες. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8 και τροπολογία 9 υπέρ, κατά, Α, η συμβατά αλλά όχι ταυτόσημα. Τροπολογία 8 λοιπόν. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 8 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 8. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ υπέρ της τροπολογίας 9. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 9 παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 καταπίπτει. Και συνεχίζουμε με την τρία της απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τέσσερα της ίδιας επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου, οι διερμηνείς δεν ακούν δυστυχώς. Εάν θέλετε μπορούμε να ψηφίσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Έμπλ 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Has everybody voted? Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε λοιπόν με το σημείο 13. Τροπολογίες 1 και 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 3 καταπίπτει, ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αποφάσεως απαλλαγής, άρχεται η ψηφοφορία. Δεν συμμετέχουν όλοι οι βουλευτές. Παρακαλώ ψηφίστε αν θέλετε γιατί θα κλείσω την ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας λοιπόν. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του κλεισίματος των λογαριασμών. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. <coughs> Ψήφισμα. Συμβεβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι τροπολογίες 7 έως 10 εκπίπτουν. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 11. Υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας 11. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε Τροπολογία 11. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεν ψηφίζουμε τις τροπολογίες της ΛΥΜΠΕ 1, 2, 3, ΛΥΜΠΕ 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. Συνεχίζουμε το σημείο 14, τροπολογίες 1 και 2, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται τροπολογία 3 εκπίπτει ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αποφάσεως ε, περί απαλλαγής. Ε, άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται κλείσιμο λογαριασμών, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, βεβαίως. Τροπολογία 10, λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11, υπέρ κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση από της τροπολογίας 11, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ της 14. Κατά. Α, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 12. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία 12. Υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας 12. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 14. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές και. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Τροπολογία 18 ηλεκτρονική ψηφοφορία. ηλεκτρονική επαλήθευση, λοιπόν, ολοκληρώθηκε, εγκρίθηκε. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Τροπολογία 23 να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ο, πέρας της ψηφοφορίας. μεγάλη διαφορά εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω πως έχει εγκριθεί, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Η τροπολογία 25, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. <coughs> Πέρασε εγκρίνεται. Η 26 εκπίπτει, συνεχίζουμε με την τροπολογία 27, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 28, κατά τμήματα η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση επί του πρώτου τμήματος της τροπολογίας 28. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Was rejected, Second part. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 29, τι σημαίνει ότι η 29 καλύπτεται από την 30. Σημαίνει ότι Α, ε, με την 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επομένως η 3 εκπίπτει. Τροπολογία 31 υπέρ. Υπέρ της 31. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 32 εκπίπτει. Τροπολογία 33 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Υπέρ της 35. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 35. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Η τροπολογία 35 εγκρίνεται. 36 υπέρ. 36 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 36. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 39. Αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ε, στην τροπολογία 1 των μεταφορών υπέρ κατά θείο των μεταφορών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με το σημείο 15. Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Τροπολογία 1. Τροπολογία 1, παράγραφος 1, υπέρ, κατά, αποχέσε, απερίφθη. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της προτάσεως απαλλαγής άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο των λογαριασμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με το ψήφισμα. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Έκον 1 είναι εκτός πεδίου. Θα το ψηφίσουμε. Θα το ψηφίσουμε. Υπέρ της έκον 1 κατά αποχές απερίφθη. Έκον 7 υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Σημείο 16. Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. τροπολογίες 1 και 2, πρόταση για τη χωρίς απαλλαγής υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απαλλαγή αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Για το κλείσιμο λογαριασμό ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Το σχέδιο ψηφίσματο. υπέρ. Τροπολογία 7 κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές και χρειάζεται ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 8 και τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. NV2 είναι εκτό πεδίου εφαρμογή, αλλά θα πρέπει να την ψηφίσουμε. Ψήφι υπέρ τη 2 τη επιτροπή περιβάλλοντο Περιβάλλοντος, κατά αποχές, απορρίπτεται. MV3 πρώτο τμήμα έχει καλυφθεί το δεύτερο ως προσθήκη. Ψηφίζουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά απόχε. εγκρίνεται. Η 7 τη επιτροπή περιβάλλοντο υπέρ κατά αποχές, δεν είναι σαφέ. ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ, επαλήθευσης. Αρχίζει τώρα. Πέρας. Α, όχι, σαν δεν ήταν σαφέστατο, συγγνώμη. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματο. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε το σημείο 7, Ευρωπαϊκό, 17, συγγνώμη, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων. Η τροπολογία είναι υπέρ κατά, απόχες εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα αρχίζει για το σύνολο. Vote It's a top. Πέρας εγκρίνεται. Συνεχίζουμε ηλεκτρονική για το κλείσιμο των λογαριασμών. Electronic vote Αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Electronic vote is closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος, τροπολογία 7, υπέρ, κατά, άποχες, δεν είναι σαφές. Και θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τροπολογία 17. Α, συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρο. 7. Η τροπολογία υπαριθμών 7. Ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 8. Ψήφι Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 9. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο NV4 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίζουμε την 4 ε, της NV, είναι βέβαια εκτός πεδίου εφαρμογής, αλλά ηλεκτρονικά θα την Ψήφισατε όλοι. Πέρα. Απέριπτ. MV7 Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος, ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχίζει τώρα. Πέρας προτρέχω κάθε φορά. Ε, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα θα πάμε στο σημείο 18. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Η τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Ας το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Χρειάζεται ξανά να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ναι, ναι. Το σύνολο της απόφασης απαλλαγής πρέπει να... Now we vote on postponement. Α, τώρα θα ψηφίσουμε για την αναβολή. Όσοι ψηφίζουν υπέρ είναι υπέρ της αναβολής, προσοχή. Όσοι ψηφίζουν κατά ε, θέλουν να χορηγηθεί η απαλλαγή. Λοιπόν, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Άρα υπερψηφίστηκε η αναβολή. Τώρα για το κλείσιμο των λογαριασμών. Uh-huh. We vote electronically on the, on the, uh, Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε για το κλείσιμο των λογαριασμών. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο των λογαριασμών. Mm. Mm. Okay. Here we have the same. If you vote... Λοιπόν, και εδώ ισχύουν τα ίδια. Αν υπερψηφίσετε, είστε υπέρ της αναβολής. Αν καταψηφίσετε, θέλετε να κλείσουν οι λογαριασμοί. Επαναλαμβάνω. Όσοι ψηφίζετε υπέρ, σημαίνει ότι είστε υπέρ Τη αναβολή του κλεισίματο των λογαριασμών. Αν καταψηφίσετε, θέλετε να κλείσουν οι λογαριασμοί τώρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. So it's 14 uh, in favor of... 14 υπέρ της αναβολής. Τώρα ερχόμαστε στο σχέδιο ψηφίσματος, στην τροπολογία 8. Ψήφι κατά άποχες απορρίπτεται. Η τροπολογία υπερθμόνα ναι, Κατά αποχές απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. Παρακαλώ. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 10 ηλεκτρονικά. Δηλαδή 9 διορθώνει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, Κάρμεν. Αρχίζουμε λοιπόν την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ΕΝΕ. Πέρασε. Ε, απορρίπτεται σαφώς. τροπολογία 10. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Θέλετε έλεγχο για την 11, ηλεκτρονική επαλήθευση, ωραία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Check is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ, ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 13. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας δεν κρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 14 Επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 Επέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 16 πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Ελέγχουμε τη 18 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Η τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν την 20. αποχές. Αν κρίνεται, σαφές. το απολογή 21. Είκοσι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα, ψηφοφορία κατά τμήματα του αρχικού κειμένου. Τμήμα πρώτον, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος, παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα του αρχικού κειμένου. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Electronic check is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογικό 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. LV2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε για την MV2. Ωραία. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία και αν ψηφίσατε όλοι, τελειώνει. Απορρίπτεται. Η τρία της ΕΝΒΗ υπέρ Τροπολογίες τρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος κατά αποχές εγκρίνεται. ΕΝΒΗ τέσσερα εκτός πεδίου εφαρμογή, αλλά την ψηφίζουμε παρόλα αυτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΕΝΒΗ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, τελική ψηφοφορία, παρακαλώ. Η κυρία Γιάλα, στην παράγραφο 6, εγκρίναμε την τροπολογία 20, έτσι δεν είναι. Μάλιστα, της κυρίας Ανδρέασεν. Και μετά, τροπολογήσαμε την ίδια την παράγραφο. Γιατί ψηφίσαμε το αρχικό κείμενο αλλά υπερψηφίστηκε και τροπολογία. Εκεί κάτι τρέχει. Ναι, όντως, υπερψηφίσαμε την 20, καταψηφίσαμε την 21. Ναι, και το αρχικό κείμενο τι έγινε, δεν υπήρχε αρχικό, αφού ήδη είχε τροποποιηθεί με την 20. Το έχει ελέγξει η γραμματεία και η ψηφοφορία κατά τμήματα θα είχε καταπέσει μόνο εφόσον είχε εγκριθεί 21, αλλά 21 σαφώς απερίφθη. Άρα χρειάστηκε να κάνουμε την ψηφοφορία κατά τμήματα και βγάλαμε τη λέξη Αλλά Αυτό ήταν που πέρασε κατά πλειοψηφία. Είναι σαφή τα πράγματα. Ναι, λέει η κυρία Γιάλα, αλλά είπαμε το αρχικό κείμενο δεν ήταν πλέον αρχικό, αφού πέρασε 20 ήταν ήδη τροποποιημένο. Έχετε δίκιο, αλλά η λέξη potential δεν είχε σχέση με την τροπολογία 20. Δεν ε, θίγει. Δεν αφορούσε τη λέξη potential που βγήκε η τροπολογία 20. Άρα μπορούσαμε και να το ψηφίσουμε και να το βγάλουμε όπως και έγινε κατά πλειοψηφία. Αν αυτό δεν ισχύει, στη διάθεσή σας να μας πείσετε, αλλά η γραμματεία είναι πολύ σίγουρη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα το ψηφίσαμε και η πλειοψηφία της Επιτροπής αποφάσισε, δεν θυμάμαι, 14 προς κάτι, εν Καλώ Καλώς, καλώς. Ο κύριος Χερμπράντη, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή μας ότι εγκρίνοντας την τροπολογία 14 και 16 επί της ε, μπαίνουμε στην ουσία μάλλον της έρευνας της Όλαφ και ε, διατρέχουμε τον κίνδυνο να ε, εγκρίνουμε πραγματικά περιστατικά εσφαλμένα. Ε, σύμφωνα με την προφόρηση που έχω εγώ ως εισηγητής Όλαφ, ε, δεν ερευνά τη σύμβαση SNA Φίλιο. Τώρα έχουμε βάλει ε, το θέμα αυτό στο ψήφισμα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Σας προειδοποιώ όμως ότι υπερψηφίζοντας το, το, το ψήφισμα υιοθετούμε κάποια λανθασμένα στοιχεία που δεν ευσταθούν και παρακαλώ να καταψηφίσετε το ψήφισμα. Μάλιστα, αυτή ήταν η σύσταση του εισηγητού. Ποιο θέλει το λόγο για διαδικαστικό, ζητάτε το λόγο. Ο κύριος Σάβαρμα. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να ενημερώσω την Επιτροπή εξ του ΕΛΚ γιατί θέλουμε να αναβάλουμε την απαλλαγή απλούστατα γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η αμφισημία, η ασάφεια και ε, ε, τα σκοτεινά σημεία για ε, τη θέση της γυναικής διευθύντριας. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε εδώ και όπως είπε προηγουμένως και ο εισηγητής, ε, ενώ αρχίζουμε να ψηφίζουμε, έχει γίνει πολύ παρασκηνιακή δουλειά. Και παρακαλώ να μην δώσουμε απαλλαγή σε έναν οργανισμό ε, όπου επικρατούν ζώνες. Και σε ό,τι αφορά τα σχόλια του εισηγητού τώρα μόλις, αυτό τώρα είναι φιλοσοφική συζήτηση. Ας μην μπούμε τώρα σε αυτά τα χωράφια. Όταν ψηφίζουμε τροπολογίες που περιλαμβάνουν ένα κείμενο που μπορεί να συνδέεται με τις έρευνες της Όλαφ, αυτό είναι θέση του εισηγητού. Αυτή η τραπός δεν μας οδηγεί πουθενά, παρά μόνο σε μεγαλύτερα προβλήματα. Αν συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική τροπολογίες 14 και 16, έχουν όντω ένα κείμενο που αφορά στην παραγωγή βίντεο, αλλά τι σχέση έχει αυτό με το γεγονός ότι ψηφίζουμε κατά της χορήγησης απαλλαγής. Γιατί τα αναμειγνύουμε αυτά τα δύο. Απλώς ήθελα να σας ενημερώσω γι' αυτά. Okay, that was a point of order. Διαδικαστικό ήταν αυτό. Άλλη πολιτική ομάδα θέλει το λόγο για αυτό το ζήτημα. Κάθε ομάδα, παρακαλώ, είναι σαν για άλλα σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ναι. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Γκερμπράντι. Δύο τροπολογίες είναι αυτές, η 14 και η 15 λέει η κυρία Γιάλα. Και τι λέγουν, ότι η ε, Όλαφ ερευνά κάτι το οποίο δεν ισχύει. Γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον στα σημεία ε, για τα οποία θα κλητευτεί η Διευθύντρια ε, δεν είναι σχετικά με αυτό. Αυτό θέλω από πω στον κύριο Γκέμπραντι, ότι ε, θεωρούμε δεδομένο κάτι ε, το οποίο ξέρουμε ότι δεν είναι αληθές. Τώρα λεπτομέρειες δεν ξέρουμε, αλλά αυτό θα το θέσουμε υπόψη και τις διευθύντριες της του Ευρωπαϊκού Αυτού Οργανισμού. Ναι, είμαστε στην ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρο. Θα δώσω το λόγο σε όλε τι πολιτικέ ομάδε διαδικαστικά. Υποχρεωμένοι δεν είμαστε, αλλά μπορούμε για να καθορίσουμε τη στάση μα στην ψηφοφορία. Θέλει οπωσδήποτε να μιλήσει κάθε πολιτική ομάδα ή μπορούμε να συνεχίσουμε να ψηφίζουμε. Δεν θέλει κανείς άλλος συντονιστη Ωραία. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία και ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Okay, everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Vote is closed. So that was adopted. Πέρας, εγκρίθηκε. 15-12 χωρίς αποχές. Ωραία. Προχωρούμε. Είμαστε στο σημείο 19. Κοινοτική υπηρεσία ελέγχου της αλίας. Η τροπολογία ψηφίπερ Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απόφαση χορήγησης απαλλαγής. Συνολικά αρχίζει τώρα. Και αν ψηφίσατε όλοι. Κλείνει. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο των λογαριασμών. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος, τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 είναι τεχνική διόρθωση και δεν την πληρώνουμε. Πες 1, η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΠΕΣ 2 της Επιτροπής Αλίας ε, τη ψηφίζουμε παρόλο που είναι εκτός πεδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΠΕΣ 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το ψήφισμα στο σύνολό του. Αρχίζει το ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εγκρίνεται σαφώς και συνεχίζουμε με το σημείο 20. Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων. Εύσα. Τροπολογία 1 και 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει τώρα για τη χορήγηση απαλλαγής. Πέρας. πρόταση απόφασης για το κλείσιμο λογαριασμών, ηλεκτρονική ψηφοφορία και πάλι αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Το σχέδιο ψηφίσματος, η τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 10, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία περιθμών 11. Αρχίζει τώρα. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 14 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 15 επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 16 επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει 19. 20 υπέ. κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία παρθμών 20 αρχίζει τώρα. Πες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 21 ψήφι πέ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 22 με προφορική τροπολογία την οποία βλέπετε δίπλα. Ε, είναι σχετικά με τη μετακίνηση ε, του προσωπικού της αρχής ε, σε λόμπι και σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων. Ποιος είναι υπέρ αυτής της προφορικής τροπολογίας που βλέπετε δίπλα στην 22 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αν εγκριθεί λέει 17, καταπίπτει 26. Εγκρίθηκε 17, οπότε καταπίπτει 26. 27 υπέρ κατά ελέγχουμε την 27 ηλεκτρονικά. Αρχίζει η επαλήθευση τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 28 ψηφίπε. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 28. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 30. Ε, Αρχίζει η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 31. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 32. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο για την 32. Παρακαλώ. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Όπως σας είπα. Άλλωστε. Εφόσον εγκριθεί 32 καταπίφθη 33 αλλά περίφθη 32 οπότε ψηφίζουμε την 33. Ψηφί πέ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Λοιπόν, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία υπαριθμών 34. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Αγκρίνεται. 35 ψήφι υπέρ. Τις 35. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την 35 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Παραμένει ανοιχτή η ψηφοφορία για να ψηφίσετε. Τώρα κλείνει. Απορρίπτεται. Η 36 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 είπε. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Διότι δεν σηκώνετε χέρια μερικοί. Άρα χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος που αρχίζει τώρα. Vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV4 Υπέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. MV5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το σύνολο του ψηφίσματος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Παραμένει ανοιχτή αν θέλει κάποιος να ψηφίσει ακόμα. Και τώρα κλείνει. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Σημείο 21. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Τροπολογίε 1 και 2. Ψηφιπέ. Κατά. απόχέ εγκρίνονται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την απαλλαγή συνολικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Και για τον κλείσιμο λογαριασμών επίσης ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 7. Ε, τροπολογία επί του ψηφίσματος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 10. Ταυτόσημη με ποια όμως. Α, με την 11. Ωραία, τις ψηφίζουμε μαζί τότε. 10 και 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αν εγκριθούν λοιπόν αυτές οι δύο, οι 12, 13 και επόμενοι χωριστοί καταπίπτουν. Πάμε στις τροπολογίες Επιτροπής Γυναικών. ΦΑΜ 3. Υπέρ, κατά, άποχες, ε, εγκρίνεται. ΦΑΜ 8. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. ΦΑΜ 9. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. ΦΑΜ 10. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. ΦΑΜ 11. Εκτός πεδίου, αλλά ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Για την 11 της ε, Επιτροπής Γυναικών. Vote is closed. φέστατα απερίφθη. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο του σχέδιου ψηφίσματος. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. κρίνεται. Συνεχίζουμε. σημείο 22. Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Η τροπολογία ένα ζητή ε, αναβολή της απαλλαγής. Ποιος είναι υπέρ της απολογίας κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για να δοθεί η απαλλαγή, αν θέλετε να δοθεί η απαλλαγή ψηφίζετε υπέρ, αν θέλετε αναβολή ψηφίζετε κατά. Ψηφίσατε όλοι. Είπαμε το υπέρ σημαίνει ότι θέλουμε απαλλαγή, τη χορηγούμε, εντάξει, ωραία. Πάμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρώτα κλείσιμα με λογαριασμών, ηλεκτρονική ψηφοφορία και πάλι αρχίζει τώρα. Συνεχίζουμε. Πρόταση ψηφίσματος. Η τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 1. Εκτός πεδίου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4 της οικονομικής και νομισματικής υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εκόν 10, εκτός πεδίου βέβαια, αλλά την ψηφίζουμε, ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται. Εκόν 12, υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκόν 13, υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημαίνει 23. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Η τροπολογία υπερθμών 1. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα και αρχίζει η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το κλείσιμο των λογαριασμών. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται το σχέδιο ψηφίσματος και πάλι ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε σημείο 4 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Τροπολογίες 1 και 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την χορήγηση απαλλαγής. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Και τελειώνει. Εγκρίνεται. Το κλείσιμο λογαριασμό, ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με το σχέδιο ψηφίσματος. Έχουμε την τροπολογία παριθμών 8, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Νέα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, ηλεκτρονικός έλεγχος για την ε, τροπολογία 9, αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας.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 Ψηφίσατε όλοι. Βεβαίως. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίψετε. Η τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές. Έχουμε ηλεκτρονικά τη 16. Αρχίζει η πολίτευση.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 κατά αποχές εγκρίνεται. NV2 εκτός πεδίου αλλά την ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 5 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV10 ως προσθήκη όμως υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, η πρόταση ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε στο σύνολό της αρχίζει του ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε. Σημείο 25. Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Οι τροπολογίες 1 και 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την πρόταση συνολικά για την απαλλαγή. Αρχίζει τώρα. Ψήφισετε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το κλείσιμο των λογαριασμών, ηλεκτρονική και πάλι ψηφοφορία αρχίζει τώρα.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 υπέρ, όχι υπέρ, ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας. κρίνετε. Σημείο 26. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, η ΕΜΣΑ. Οι 1 και 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για την απαλλαγή αρχίζει τώρα. Everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Για το κλείσιμο του λογαριασμού ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Συνεχίζουμε με ε, την πρόταση ψηφίσματος. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 10 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικά δεν είναι σαφές. Vote is Πέρας προφορίες και εγκρίνεται. Αν εγκριθεί 10 κατά 11 και προχωρούμε, τραν 2 υπέρ της 2 της Επιτροπής Μεταφορών κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα, 4 τη τραν εκτός πεδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 6 και πάλι εκτό πεδίου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος αρχίζει τώρα. Και ψηφίσατε όλοι. Τελειώνει. Εγκρίνεται. Ακολουθεί το θέμα 27. Ευρωπαϊκός Αγωνισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ΕΝΙΣΑ. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στο σύνολό της η πρόταση αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο λογαριασμών. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Πρόταση ψηφίσματος. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική, η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σύνολο του ψηφίσματος. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. 28. Σιδηροδρόμων. Τροπολογία 1 και 2 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνονται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του, ε, της προτάσεως. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Κλείσιμο λογαριασμών, ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζω πρόταση ψηφίσματος. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται αυτή. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 2 out of scope υπέρ. Κατά. Αποχές αυτή απορρίπτεται. Τραν 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 29. Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Αγορών και Χρεογράφων. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σύνολο της προτάσεως. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρασε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο λογαριασμών. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Πρόταση ψηφίσματος, τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκον 1, out of scope, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έκον 10, out of scope, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται και αυτή. Έκον 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και έκον 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σύνολο της προτάσεως ψηφίσματος. Τέλος. Εγκρίνεται. Το υπαριθμόν 30. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Εκπαιδεύσεως. ETF. Τροπολογίες 1 και 2 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνονται. Πρόταση στο σύνολό τη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Κλείσιμο λογαριασμών. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Απασχόλησης 2 out of scope υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 out of scope υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της προτάσεως ψηφίσματος. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συνεχίζω. Θέμα 31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Τροπολογίες 1 και 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Ηλεκτρονική ψήφος αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Κρίσιμο λογαριασμών. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Τέλος. Πρόταση ψηφίσματος, τροπολογία 7, υπέρ, κατά αποχές, Ας επαληθεύσουμε. Τροπολογία 7. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε. Θαυμάσια. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 9. Ψηφίσατε. Θαυμάσια. τέλο. Εγκρίνεται. Έμπλ 1. Οτοσκόπ υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Έμπλ 6. Οτοσκόπ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Ακολουθεί το υπαριθμό 32. Ευρατόμ Supply Agency. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απόφαση στο σύνολό της. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα για τους λογαριασμούς, για το κρίσιμο των λογαριασμών. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Πρόταση ψηφίσματος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία που αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. 33. Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης. Καλό θέμα αυτό. για την Επιτροπή μας working and living conditions χωρίς διάλειμμα. Λοιπόν, ε, τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Κλείσιμο λογαριασμών. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει. Ψηφίσατε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Συνεχίζομαι. Πρόταση ψηφίσματος. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 3. Ψηφίσατε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές πάλι. Παρακαλώ, ενεργότερη συμμετοχή. Αρχίζει πάλι η, αρχίζει μάλλον η ψηφοφορία, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ψηφίσατε. Τέλος. Σαφώς εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές πάλι. Νομίζω ότι εγκρίνεται ηλεκτρονική ψήφος. Τροπολογία 5 λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται σαφώς. Και συνεχίζουμε. Ample 1, out of scope. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ample 2, out of scope. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται και αυτή. Στο σύνολο του το ψήφισμα, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. 34. Τροπολογίες 1 και 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Τέλος. Εγκρίθηκε. Κλείσιμο λογαριασμών αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται και αυτή πρόταση ψηφίσματος, τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, με συγχωρείτε, κατά, λέει ο πρόεδρος πάλι, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφέ. Το αποτέλεσμα ηλεκτρονική ψήφος τροπολογία 10. Ψηφίσατε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά εποχές Κρίνεται. Α, επαλήθευση έχει καλώς. Για την 14 αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Συνεχίζω. Λίμπε 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8. Αοντοσκόπ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του, η ηλεκτρονική ψήφος, πέρας, εγκρίνεται. 35 Ευρωπόλ. Τροπολογίες 1 και 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η ηλεκτρονική ψήφος αρχίζει. Ψηφίσατε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται ηλεκτρονική ψήφος για το κλείσιμο λογαριασμών. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Πρόταση ψηφίσματος. Τροπολογία 7. Υπέρ. Α, με συγχωρείτε, έχει αποσυρθεί. 8 επίση έχει αποσυρθεί. Ναι, και η 8. Άρα, δεν Γίνεται τη ψηφοφορία. Α, ναι, αλλά έχει αποσυρθεί όμως, αλλά θα γίνει χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 8. Ορθώς, ναι. Καλά λοιπόν. Ξεχωριστή ψηφοφορία για την 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σωστό. Α, επαλήθευση λοιπόν. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 13 εκπίπτει εφόσον έχει εγκριθεί η 10, έτσι δεν είναι. Σωστά. Τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι οι περισσότεροι απέχουν. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για την τροπολογία 15. Αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Ορίστε κύριε Σάπαρμα. Η 14 είναι κρίθη. Αν θέλετε παρήθευση. 14. Ηλεκτρονική ψήφος για τη 14. Η ηλεκτρονική Ψήφό για την 14, τροπολογία 14. Τέλος. Μου είχε φανεί σαφές το αποτέλεσμα, αλλά εφόσον ζητείτε ηλεκτρονική ψήφο, βέβαια το αποτέλεσμα είναι ακόμα σαφέστερο. Τι να κάνω, δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα. Τώρα, η 16. Υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε και εδώ 16 αρχίζει πέρας ψήφισατε όλοι λοιπόν εγκρίνεται 17 υπάρχει και προφορική τροπολογία εδώ ο κύριος Σάβαμα έχει ως εξή. Τροπολογία 17. Από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου σημειώνει ότι το γραφείο μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες προσλήψεως και ζητεί να διευκρινιστούν ενδεχόμενες ελλείψεις σε σχέση με τις διαδικασίες προσλήψεως. Ορισμένες από τις διατάξεις του καταστατικού των υπαλλήλων ενδέχεται να αποτελούν ή να προκαλούν σημαντικό γραφειοκρατική, σημαντική γραφειοκρατική επιβάρυνση και το υπόλοιπο να διαγραφεί. Έχει κανείς ένσταση για την προφορική τροπολογία? Όχι, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία, δηλαδή την τροπολογία 17 με αυτή την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19. Θέλετε παρήθευση για 18. Καλά. Αρχίζει. Τέλος. Απερίφθη. 19. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ας, ας επαληθεύσουμε όμως την 20. Ψηφίσατε. Τέλος. Απερίφθη. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 7 out of scope υπέρ κατά αποχές πολύ, πολύ περιορισμένη συμμετοχή. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την ΛΥΜΠΕ 7. Τέλος. Απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σύνολο. Για το σύνολο δηλαδή. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται λοιπόν και συνεχίζουμε με το 36. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ένα και δύο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο λογαριασμών. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Πρόταση ψηφίσματος. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Εφόσον εγκρίνεται η 9, εκπίπτουν οι 10 και 11. Συνεχίζουμε τη 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Επαλήθευση για την 12. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. Εφόσον όμω εγκρίνεται η 12, εκπίπτουν 13 και 14 και συνεχίζουμε με την 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές, παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση, αρχίζει, Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Εκπίπτει. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε με το σημείο 37, Frontex, τροπολογίες 1 και 2, υπέρ, κατά, αποχέσε, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο των λογαριασμών. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με το ψήφισμα. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 10. Η ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν τροπολογία 10 άρχεται. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 14. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Εκτός πεδίου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 17. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθη. Λίμπε 6 εκτός πεδίου υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Το ψήφισμα στο σύνολό του με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Vote is It's adopted. Συνεχίζουμε με το σημείο 38 Ευρωπαϊκή Αρχή GNSS. Είναι η υποπτική αρχή GNSS. Τροπολογίες 1 και 2 υπέρα. Κατά αποχές. Εγκρίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται κλείσιμο λογαριασμών, ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία. Πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με το ψήφισμα. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχέσε απερίφθη. Το σύνολο του ψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα ε, με τις επιχειρήσεις. Κοινέ επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Okay. Discharge for 2011 Artemis Embedded Computing Artemis ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών. Τροπολογία 1 και τροπολογία 2 λέει ο πρόεδρος. Οι τροπολογία 1, 3 και 5 είναι ταυτόσιμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κλείσιμο λογαριασμών, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με το ψήφισμα. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 12 Everybody voted. ψήφισαν όλοι πέρασε. απερίφθη Επομένως ψηφίζουμε την τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Η ηλεκτρονική επαλήθευση τη τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 11. Προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. ζητά από την Επιτροπή να ε, πληροφορήσει την ε, αρχή απαλλαγή όσον αφορά την νομιμότητα της καταστάσεως όσο γίνεται ε, το συντομότερο δυνατόν υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται στο ψήφισμα, το ψήφισμα στο σύνολό του, η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε λοιπόν με το σημείο 40, Clean Sky, αεροναυτική και περιβάλλον. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο των λογαριασμών υπέρ. Ψήφισαν όλοι, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 ε, υπέρ κατά αποχές ε, ψηφίζεται 10 ε, το ίδιο, 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος ε, άρχεται πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στο 41 ΕΝΙΑΚ, ηλεκτρονικός αριθμητικός ολοκληρωτής και υπολογιστής. Τροπολογίες 1-4-5 ταυτόσιμες ταυτόσμες υπερ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπο, ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο των λογαριασμών. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρόταση ψηφίσματος. Τροπολογία 6 και 8. Αυτές είναι ταυτόσιμες υπέρα. Κατά. δεν είναι ταυτόσιμες. Ο εισηγητής παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, στο ψήφισμα ξεκινάμε με την τροπολογία 9. Ναι, ναι, ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος. Ευχαριστώ κύριε εισηγητά. Λοιπόν, μετά από τρεις ώρες έχει επέλθει μία κόπωση. Ξεκινάμε λοιπόν με την τροπολογία του Πολ Ρούμπιχ, τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Τροπολογίες Γεμπράντι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του εισηγητού ζητά από την Επιτροπή να πληροφορήσει τις αρχές, την αρχή απαλλαγής σχετικά με την νομιμότητα της καταστάσεως. Το συντομότερο δυνατό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πολ Ρούμπιχ, τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 είναι Σαγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου του ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με κυψέλες καυσίμου και ε, ε κυψέλες υδρογόνου, FCH, τροπολογίες 1-3-5, ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κλείσιμο των λογαριασμών. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται για το κλείσιμο. Συνεχίζουμε με το ψήφισμα. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε η ηλεκτρονική επαλήθευση για το 9. Α, να ψηφίσουμε on block. Ωραία. Από κοινού λοιπόν υπάρχει κάποιος που αντιτίθεται στην ψηφοφορία από κοινού. Όχι, 9 με 11 μπλοκ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται επί του ψηφίσματος στο σύνολό του, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Σημείο 43. Ε, καινοτόμων φαρμάκων. IMI 1 μέχρι 5 ταυτός με υπερκατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία ηλεκτρονική ψηφοφορία κάτι δεν λειτουργεί εδώ Α, τώρα άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Κλείσιμο λογαριασμών, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Συνεχίζουμε με το ψήφισμα. Τροπολογία 9 Ε, ε, συμφωνείτε από την τροπολογία 9 μέχρι 15 αν μπλοκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου του ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Πολύ ωραία. Κοινή επιχείρηση για τον ΙΤΕΡ 1-3 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα έχει περατωθεί. Εγκρίνεται. Κλείσιμο λογαριασμών, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 9 για το ψήφισμα υπέρ, κατά, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 9 του ψηφίσματος. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με το σημείο 45. Κοινή επιχείρηση Σέζαρ. 1-2 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με το κλείσιμο των λογαριασμών. Ηλεκτρονική ψηφοφορία πάντα. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε τώρα με το ψήφισμα Τροπολογία τραν 3. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του Uh, Μια ερώτηση προς την Επιτροπή θα απευθύνω τώρα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ψηφοφορίες πρώτα. Λοιπόν, η επιχείρηση Σέζαρ ε, έχει υπερψηφιστεί με σαφή πλειοψηφία. Τώρα κοιτάξτε, ο κύριος υπουργό είναι εδώ και αναμένει, επομένως προτείνω, προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία για τα άλλα όργανα, να κάνουμε τις ψηφοφορίες αυτές το απόγευμα. μαρτυρίες, όχι, να συνεχίσουμε. εντάξει. Συνεχίζουμε, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόταση απαλλαγής για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Okay. 1. Τροπολογία 1. Υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας 1. Κατά. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 2 και τροπολογία 4. 2 και 4. Υπέρ. Υπέρ. Κατά Ε, αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ. Τροπολογία 5, είμαστε στο ψήφισμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ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 11 ψήφοι υπέρ, 16 κατά, περίφθη. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Όχι, έχει καταπέσει, συγγνώμη, 23 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία που έχει ζητήσει το ΕΛΚΑ ε, για την 24. Κύριε Κάλφιν, ε, θα ήθελα να αποσύρω την τροπολογία αυτή, λέει ο κύριος Κάλφιν. Θα ήθελα να αποσύρω την τροπολογία 24, λέει ο κύριος Κάλφιν. Εντάξει, επομένως απεσύρθη τροπολογία 25 υπέρ. Κατά υπέρ, υπέρ της 25, υπέρ της 25, κατά της 25, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 29 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. Ψηφίζουμε την τροποποιηθή, το τροποποιηθέν ε, ψήφισμα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Υπερψηφίστηκε και συνεχίζουμε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τροπολογία 1, υπέρ της τροπολογίας 1, κατά, αποχές, απερίφθη, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εδώ δεν υπάρχουν λογαριασμοί. Πέρας της ε, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ενεκρίθη. Τροπολογία 2 του ψηφίσματος υπέρ, κατά, Απόχες, απερίφθη. Τροπολογία 1 της ΑΦΕΤ έχει καλυφθεί από την τροπολογία 2, αλλά η τροπολογία 2 απερίφθη. Από τη στιγμή που η τροπολογία 2 δεν εγκρίθηκε, πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 1 της ΑΦΕΤ υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονική ε, επαλήθευση από τις τροπολογίες 1 της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων άρχεται πέρας απερίφθη. Τροπολογία 3. Υπέρ της τροπολογίας 3. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 καλύπτεται από την 8, τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 και 12 συνδυασμένες σε, μια νέα, σε ένα νέο κείμενο, το οποίο είναι γραπτό, το έχετε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 13 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση του επί της 14 υπέρ, ε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 άφετ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία για τη 15. Υπέρ, υπέρ της τροπολογίας 15. Σηκώστε τα χέρια σας. 15. Είναι σαφές ότι εγκρίνεται τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 άφετ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 21. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές ε, δεν είναι σαφές τροπολογία 28 ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Επομένως, οι τροπολογίες 29, 30 και 31 εκπίπτουν. Τροπολογία 5 της άφετη πέρα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία από τις τροπολογίες 32. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 33. 33 μέχρι 38 μπορούμε να τις ψηφίσουμε on block. Πολύ ωραία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική ε, ψηφοφορία. 33 με 38 ψηφίζουμε on block τις τροπολογίες αυτές. Πέρας της ψηφοφορίας. Ισοψηφία επομένως απορρίπτονται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 42. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Τροπολογία 40, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, δεν είπα ποιο είναι το αποτέλεσμα, γιατί δεν είδα το αποτέλεσμα, λέει ο Πρόεδρος της προηγούμενης τροπολογίας. 14 ε, ισοψηφία και απερίφθη λοιπόν. Α, για την η τροπολογία 42 απερίφθη. Ναι. Τώρα να ψηφίσουμε τη 40 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 40. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση για την ε, τροπολογία 43. Πέρας. Ισοψηφία, επομένως απορρίπτεται. Τροπολογία 44, υπέρ, κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές ε, απε, <coughs> συγγνώμη απερίφθη τροπολογία 8 άφετ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Συμβιβαστική τροπολογία 3 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. It's adopted. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, Ξέχασα όμως τη 48 και ζητώ συγγνώμη. Επανέρχομαι. Ψήφι υπέρ τη 48. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε τη 48. Μάλιστα, αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές Έλεγχος, παρακαλώ, ηλεκτρονικός. Check is open. Everybody voted. Check is closed. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. It's rejected. 53. Απορρίπτεται. Η 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 53. Check is closed. It's rejected. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 5 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος της 9 της Επιτροπής Εξωτερικών. Αρχίζει τώρα η επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 αφέτ υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι σαφές και πάλι. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει τώρα. Everybody voted. Vote is... Ε, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. It's adopted. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 6. Ψηφί υπέρ. Τη συμβαστικής τροπολογία παριθμών 6 κατά αποχέ. δεν είναι σαφέ. Σας παρακαλώ. Συμβαστική 6. Ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Vote is closed. Πέρας. Α, αγκρίθηκε σαφω. Η τροπολογία 7 ψήφι. Υπέρ παρακαλώ. τη επιτροπή Εξωτερικών. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά παρακαλώ αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 64 ψήφι υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 64. Πέρας. Απορρίπτεται. απολογία 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί την 66 αρχίζει τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές παρακαλώ ηλεκτρονικά ελέγχουμε την 68 für die nur Frau Kressel kann ich umdrehen. Nur we can't just leave him in front of the door. Ja, Yeah, machen wir das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 70 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το σύνολο τώρα. Αρχής ψηφοφορία. Load is closed. Πέρας. Ωραία. Και τώρα δεύτερη απόπειρα. Δεν μπορούμε να, αφήσουμε, να αφήνουμε τον Υπουργό, τον Ρουμάνο, τον οποίο εμείς προσκαλέσαμε, να περιμένει. Λοιπόν, δύο τι να έχουμε τώρα. Είτε θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία και να επανέλθει ο Υπουργός στις 3 το απόγευμα, είτε θα του δώσουμε την ευκαιρία τώρα να μιλήσει, να ανταλλάξουμε απόψεις και να αναβάλουμε τις υπόλοιπες ψηφοφορίες για την απογευματινή συνεδρίαση. Να ψηφίσουμε και γι' αυτό. Ποιο είναι υπέρ τη αναβολή των ψηφοφοριών. Παρακαλώ κύριε Γκρέσλα. Μα είναι θέμα ευγενία. Τον έχουμε προσκαλέσει για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και θα πρέπει να τον δεχθούμε την ώρα που τον καλέσαμε. Λέω εγώ τώρα. Ναι, είναι θέμα ευγένεια. Όταν καλείς κάποιον, ο υπουργό επέδειξε μια ευελιξία, μα πρότεινε να έρθει στι 3. So Και το κοινοβούλιο είναι κυρίαρχο και μπορεί να αποφασίσει. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ της αναβολής των ψηφοφοριών για την απογευματινή συνεδρίαση. Για να δούμε τώρα τον Υπουργό. Λοιπόν, συνέχιση των ψηφοφοριών στις 3 η ώρα το απόγευμα. Ποιος είναι υπέρ της αναβολής. Κατά. Και η ηλεκτρονική επαλήθευση τώρα για την αναβολή. Αρχίζει τώρα. Okay, vote is closed. Πέρας. <laughs> okay. Uh -huh. Okay, so we, we invite the minister... Λοιπόν, α, θα δούμε τον Υπουργό το απόγευμα. Απερίφθη η πρόταση αναβολής των ψηφοφοριών. Okay, sorry, sorry, sorry. Please stay. We have the we have the meeting room only from. Γράψτε λάθος. Η ε, αίθουσα διατίθεται από τις 4 και μετά. Άρα μία δυνατότητα έχουμε να ακούσουμε τώρα τον Υπουργό και να ψηφίσουμε στις 4. At 4 o'clock he will not be available. Ε, στις 4 δεν μπορεί ο άνθρωπος. Μα είπε ε, ότι μόνο 3 με 3,5 ε, θα μπορούσε να έρθει. Αν θέλετε να ακούσετε τον Υπουργό, τον οποίο εμείς προσκαλέσαμε, θα πρέπει τώρα να τον ακούσουμε και να αναβάλουμε τις ψηφοφορίες για τις 4 ώρα το απόγευμα. Είναι νέα δεδομένα. Λοιπόν, αυτό τώρα ψηφίσουμε. Είμαστε υπέρ του να αναβληθούν οι υπόλοιπε ψηφοφορίε για τι 4 ώρα το απόγευμα. Κατά. Ωραία. Αυτή ήταν σαφή πλειοψηφία. Θα δούμε τώρα τον Υπουργό. Σα ευχαριστώ πολύ. Short minutes, uh, we will... κάνουμε ένα λεπτάκι διάλειμμα και μετά θα δεχτούμε τον Υπουργό. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Dear colleagues, uh, let us continue. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Καλωσορίζω στην Επιτροπή μας ε, τον Υπουργό της ε, Ρουμανικής Δημοκρατίας, κύριο Όγγεν Ορλάντο Τεοντοροβίτσι. Ελπίζω να ε, προφέρω σωστά το όνομά σας. Η διαδικασία απαλλαγής για το 2010 εντόπισε τρεις χώρες όπου τα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης των κοινοτικών πορών χωλαίνει. Ε, Τσεχική Δημοκρατία, Ιταλία και Ρουμανία. Οπότε ε, γι' αυτό καλέσαμε τις ε, αρχές των λογοκρατών να απαντήσουν. Η Τσεχική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Ρουμανίας αντέδρασαν θετικά Είδαμε τον κύριο Μύροσλαφ Ματέη στις 27 Νοεμβρίου του 2011, αναπληρωτή υπουργό, ενώ ε, χρειάστηκε να αναβληθεί η αντίστοιχη συνάντηση με τον Ρουμάνο Υπουργό γιατί είχαν εκλογές στη Ρουμανία βουλευτικές το ε, Δεκέμβριο του 2012 και τώρα έχουμε τη μεγάλη τιμή που έχουμε την ευκαιρία και να σα υποδεχόμαστε κύριε Υπουργέ για να απαντήσετε στι ερωτήσεις στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Σα καλωσορίζω. Είχαμε κάποιες ψηφοφορίε, δυστυχώ καθυστερήσαμε λίγο, αλλά τώρα θα αφιερώσουμε όλο το χρόνο και θα ήθελα καταρχάς να σας δώσω το λόγο για κάποια εισαγωγικά σχόλια λίγο λεπτών. Γνωρίζετε ε, ότι έχουν εντοπιστεί κάποιες αδυναμίες και διαβάσατε και το ψήφισμά μας για την ε, απαλλαγή και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε ε, ποιες συνέπειες και σε ποια συμπεράσματα κατέληξε η ρουμανική κυβέρνηση από τις προτάσεις μας. Σας καλωσορίζουμε θερμότατα στην Επιτροπή μας και σας δίνουμε αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα σύντομα να σας παρουσιάσω τα μέτρα που έλαβε η Ρουμανία για ενισχύσει τον μηχανισμό ελέγχου και εποπτείας για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Αρχής γενομένης από το 2012 έχει λάβει μέτρα ε, για να διορθώσει τα κακό κείμενα η Ρουμανία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τις αναθέσεις έργων τα μέτρα αυτά ελήφθησαν για να διευκρινιστούν και να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες και ευθύνες των διαφόρων δομών που συμμετέχουν στις προμήθειες δημοσίων έργων και στον έλεγχο. Υπάρχει και η Εθνική Αρχή που ρυθμίζει και ελέγχει ε, τις κρατικές προμήθειες ε, που ενσωματώθηκε στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ε, ως ε, δομές εκ των προτέρων υποστήριξης που υποστηρίζονται από την ελεκτική αρχή. Ελήφθησαν μέτρα για να εδρεωθεί η εποπτική ε, αρχή και ο ρόλος της ως απορρέει από τον αντίστοιχο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και διαθεσμική συνεργασία μεταξύ των εθνικών κρατών και των κοινοτικών αρχών ενισχύθηκε και λήφθησαν οι απαραίτητες προσπάθειες για να ε, γίνονται επαληθεύσεις και εκ των προτέρων αλλά και εκ των υστέρων. Ε, οι διαγωνισμοί και οι συμβάσεις για ε, το περιβάλλον, τους διδάτινους πόρους, τα απόβλητα και τις μεταφορές έχουν τυποποιηθεί και περαιτέρω τυποποίηση των εγγράφων των διαγωνισμών επίκειται. Είναι κάτι το οποίο σκοπεύουμε να υιοθετήσουμε. Οι ε, αρχές ε, και πάλι ελέγχουν τους διαγωνισμούς για όλες τις δαπάνες που ήδη έχουν δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, ενημερώσαμε αντιστοίχως. Τέλη του 2011 η Ρουμανία δέχτηκε επισήμως όλες τις καταποκοπήν ε, διορθώσεις που πρότειναν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια θετικά μήνυματα. Ε, βλέπουμε ήδη ε, θετικά αποτελέσματα και βελτίωση ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα έγγραφα για τους διαγωνισμούς, την προκήρυξή τους και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Επίσης, ανέλαβε η Ρουμανία να διορθώσει όλες τις δαπάνες στις διαδικασίες των κρατικών προμηθειών που ε, είχαν κινήσει πριν τον Οκτώβριο του 2011. Για αυτά τα προγράμματα, η στοιχεία των προγραμμάτων που ε, μας ε, έκανε συστάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οριζόντιες εργάσιες διορθώσεις, επίσης το δεχτήκαμε θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα των δημοσίων διαγωνισμών και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της διαπλοκής και της σύγκρουσης συμφερόντων με τρόπο συστηματικό. Η ρουμανική νομοθεσία ε, είναι πολύ αυστηρή πλέον ε, για την ταυτοποίηση και καταπολέμηση της σύγκρουσης συμφερόντων με αντίστοιχες κυρώσεις και μέτρα. Έχουν ληφθεί πέρυσι στην κατεύθυνση αυτή συγκεκριμένα μέτρα που δείχνουν ότι είναι πλήρω προσιλωμένε οι ρουμανικέ αρχές στο σεβασμό ε, του ε, προγράμματος της κείμενης ε, νομοθεσίας και στη διαδικαστική αλλά και στην επιχειρησιακή φάση. Έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός και το συζητούμε με τις ελεγκτικές υπηρεσίες ακόμα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Οικονομικού Ελέγχου και ε, για όλα τα προγράμματα ε, υπάρχει μια εκτίμηση κινδύνου για να εντοπίσουμε ε, κάποιες ύποπτες περιπτώσεις για απάτη, συγκρούσεις συμφερόντων, για να βελτιωθούν οι έλεγχοι στις κρατικές προμήθειες. Όλες οι διαχειριστικές αρχές έχουν ε, αναλάβει αυτή την προσπάθεια και ελέγχουν ε, τους δείκτες διαφθοράς απάτης ή σύγκρουση συμφερόντων. Έχουμε υπογράψει αντίστοιχα πρωτόκολλα με τις εθνικές αρχές, ε, με το εμπορικό μητρό για να κάνουν και οι ίδιοι ε, τους ελέγχους τους με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, με συγκεκριμένα ε, στοιχεία και βάσεις δεδομένων των θεσμικών οργάνων, πάντα σε ό,τι αφορά την ε, καταπολέμηση της διαπλοκής της σύγκρουσης συμφερόντων και της απάτης. Τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται έτσι ώστε οι αρμόδιες εθνικές αρχές να κάνουν έρευνες που είναι η Εθνική Αρχή Ακαιρεότητας Θεσμικέ συνεργασίες, ακόμα και το τμήμα πολέμηση τη Απάτη. Επιπλέον, ε, σε σχέση με την κείμενη εθνική νομοθεσία, ε, Μπορείτε να διαβάσετε λίγο πιο αργά, λέει ο Πρόεδρος, ναι. Ε, σύμφωνα, λέγω, με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις, η ε, πιστοποιητική αρχή στις δηλώσεις που κάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις Δαπάνες δεν υπολογίζει τις δαπάνες ε, που καταβάλλονται στους τελικούς αποδέκτες που είναι ύποπτοι απάτης μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή η διαχειριστική αρχή ε, κάνει όλες τις διαδικασίες μέχρι να ολοκληρωθεί το σύνολο της έρευνας. Ε, πρόσφατα έχουν ληφθεί και περαιτέρω μέτρα για να ενισχυθεί η πρόληψη σύγκρουση συμφερόντων ε, στις δημόσιες προμήθειες. Γίνονται εκ των προτέρων επαληθεύσεις πριν υπογραφούν οι συμβάσεις. Τα μέτρα αυτά όλα έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τρία επιχειρησιακά προγράμματα απαντήσαμε στις ε, επιστολές το Φεβρουάριο με τεκμηρίωση και υποστηρικτικά έγγραφα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναγνωρίζω το ρόλο της ε, πληροφόρησης ε, σε όλα τα επίπεδα για τη σύγκρουση συμφερόντων και αντίστοιχα εκπαιδεύουμε και βοηθούμε στην συνειδητοποίηση και τους υπαλλήλου που διαχειρίζονται αυτά τα προγράμματα αλλά και τους τελικούς αποδέκτες. Ε, και αναφέραμε το Φεβρουάριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις εναπομείνασες δράσεις ε, που αναφέρονται στις επιστολές της και τα μέτρα που έχουμε λάβει και σε οριζόντιο επίπεδο αλλά και ειδικά για το κάθε πρόγραμμα. Ε, είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα εκτιμήσει αναλόγως την επιτευχθήσα πρόοδο και θα προβεί σε απαραίτητες κινήσεις. Θέλω να τονίσω ότι βασικό στόχος της Ρουμανικής Κυβέρνησης είναι να καλυφθούν οι καθυστερήσεις ε, που έχουν σημειωθεί στα διορθωτικά κονδύλια και θα πρέπει ε, να αυστηρά να τηρούνται τα κριτήρια της χρηστής οικονομικής διαχείρισης για να προλαμβάνεται ε, οποιοδήποτε πρόβλημα και γι' αυτό έχουμε ε, καθορίσει και ένα αρμόδιο που θα συνεργάζεται με τις διαχειριστικές αρχές για τα ε, ευρωπαϊκά προγράμματα για να είναι πιο αποτελεσματική η διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Θα το συζητήσω και σήμερα με τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιπλέον ενημέρωση και ελπίζουμε σύντομα τα προγράμματα που έχουν διακοπεί θα συγχυστούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ποιες ερωτήσεις τυχόν έχετε. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για, τις, για την τοποθέτησή σας. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι προβλέπει η ρουμανική κυβέρνηση για την... Περιμένω λίγο μέχρι να φορέσει τα ακουστικά σας μα ενδιαφέρει, έλεγα, να μάθουμε πώς η Ρουμανική κυβέρνηση προτίθεται ή μάλλον με εφήρμοσε τις αποφάσεις διότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει προβλήματα και με την απορρόφηση των πόρων και με την υποβολή σχετικών εγγράφων. Αν μπορούσατε να μας δώσετε και αντίγραφο της ομιλίας σας, θα μπορέσουμε να το διαθέσουμε σε όλα μας τα μέλη και δια των πρακτικών. Θα αρχίσουμε τώρα με τις, υπο... με ερωτήσεις. Πρώτο ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είστε σήμερα στη διάθεσή μας για συζήτηση. Η πρόσκληση σας απευθύνθηκε μετά από δική μου πρωτοβουλία υπό την ιδιότητα του εισηγητού για την απαλλαγή του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2011. Πέρσι αρχίσαμε να συζητούμε ευθέως με τις εθνικές κυβερνήσεις διότι είχαμε διαπιστώσει ότι επανέρχεται το πρόβλημα στην κοινή διαχείριση shared management οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά την χρήση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται βέβαια και οι Ρουμάνοι πολίτε και τον ικανοποιητικό τρόπο χρήση του. Θέλαμε λοιπόν να διαφύγουμε, να ξεφύγουμε από την συζήτηση που διεξάγεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δηλαδή μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει όλες τις ευθύνες για την χρήση του προϋπολογισμού διότι συχνά διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα βρίσκονται στην βάση και δεν προχωρεί η συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις. Εδώ, στην περίπτωση αυτή, ρίξαμε το βάρος μας στα περιφερειακά ταμεία, διότι πολύ μεγάλα ποσά επιστρέφουν στις χώρες μέλη και διότι συνολικά το ποσοστό του σφάλματος μειώνεται μεν, ωστόσο σε ορισμένες χώρες μέλη διαπιστώνονται σφάλματα σε ανησυχητικά υψηλό βαθμό και αυτό ήταν και η περίπτωση της Ρουμανίας για το 2011. Χαίρο που δεχθήκατε την πρόσκληση. Ίσως η συνάντηση αυτή δεν θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα, γιατί η συζήτηση που ε, θα, γίνει με τους ευρωβουλευτές μπορεί να μην είναι πάντοτε ευχάριστη για σας. Ζητώ συγγνώμη που, όπως είπε και ο πρόεδρος μας, σας αναγκάσαμε να περιμένετε λίγο διότι καθυστέρησε λίγο η ψηφοφορία μας. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Μας περιγράψατε έναν αριθμό μέτρων που έχει λάβει η Ρουμανία για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν το 2011. Βέβαια, οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, οι διοικήσει μένουν. Γνωρίζω και υψηλού αξιωματούχου στην δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, στην Ομοσπονδιακό Κρατήριο, που λένε καμιά φορά τι με νοιάζει εμένα ποιο είναι υπουργό. Βέβαια, επισήμω, τυπικώ, την ευθύνη την φέρει η κυβέρνηση. Ωστόσο, τα διοικητικά συστήματα είναι αυτά στα οποία πρέπει να απευθυνθούμε. Μας εξηγήσατε ποια μέτρα έχετε λάβει. Εγώ συζήτησα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δω πώς κρίνει τα μέτρα αυτά, τα βήματα αυτά που κάνατε. Από όσα βλέπω, νομίζω ότι μπορώ να συναγάγω ότι ακόμη οι επιτυχίες δεν έχουν φανεί. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διακρίνει ακόμη αποτελέσματα των μέτρων που λάβατε, τουλάχιστον όχι άμεσα. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς, αντιλαμβάνομαι ότι τα μέτρα χρειάζονται κάποιο χρόνο για να αποδώσουν. Τα προβλήματα δεν διαγράφονται με μια, μια κονδυλιά, αλλά στο Υπουργείο, σας, στο υπάρχουν κάποιες προβλέψεις που θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε για το πότε δηλαδή θα αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση. Πρόεδρος, ευχαριστώ Επιθυμείτε να απαντήσετε αμέσως. Ωραία. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο ρόλος μου είναι βεβαίως να είμαι παρόν εδώ και στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν σε κάθε επίπεδο για να εξηγήσω και να παρουσιάσω τα μέτρα που έλαβε η ρουμανική κυβέρνηση για να βελτιώσει τις ελλείψεις που εντόπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2009-2011. Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο να δει κανεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βελτίωση από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνησή μας. Ωστόσο το βάρος εμείς το δίνουμε ιδιαίτερα στην διαφάνεια, διαφάνεια όλων των μέτρων. Εγώ επέμεινα και επιμένω απέναντι στην κεντρική διοίκηση στη Ρουμανία να είναι πιο διαφανής. Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα να είναι διαφανή. Εγώ επιμένω να είμαστε διαφανείς και απέναντι στο κοινό και στην Κομισιόν έτσι ώστε να μειωθεί η διαφθορά, να αποφευθούν συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε αποδίδουν. Είπα επίσης ότι δεν πρόκειται να δεχθώ συμβιβασμούς για τις συγκλούς συμφερόντων και για την διαφθορά που εντοπίζονται στα συστήματά μας. Μηδενική ανοχή λοιπόν σε τέτοια προβλήματα στη Ρουμανία. Όπως είπα, η επικοινωνία είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να μπει στο σύστημα. Όπως είπα, η κυριότητα, το ownership σε κάθε επίπεδο από τους επικεφαλείς των διαφόρων αρχών μέχρι τους υπουργούς επέμεινα όλα αυτά τα επίπεδα να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για τις αποφάσεις τους. Γιατί και η έλλειψη αποφάσεως έγκαιρα μπορεί να οδηγεί σε μεγαλύτερες ακόμα δυσκολίες από την λήψη μιας απόφασης. Εγώ επέμεινα λοιπόν ώστε να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους όλοι οι κέριοι παράγοντες. Επίσης, απλοποίηση υπάρχει χώρο για απλοποίηση του συστήματο. Εξακολουθεί να είναι περίπλοκο το σύστημα. πολλέ διαδικασίε που ίσω είναι και ένα από του λόγου που προκαλούν αυτήν την κατάσταση στη Ρουμανία. Να προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, χωρί βέβαια αυτό να αποβαίνει σε ε, βάρο τη ποιότητα και τη εφαρμογή των αρχών. Όπω τα είπα αυτά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ είμαι και ελεγκτής, auditor και στο παρελθόν έδρασα ως auditor και είμαι πεισμένος ότι χρειάζεται ένα επίπεδο απλοποίησης, αλλά όχι αυτό να αποβεί σε βάρος ενός υγιούς δημοσιονομικού συστήματος. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές αρχές στις οποίες λαμβάνουμε κάποια μέτρα και για να φανούν τα αποτελέσματα θα το δούμε και στο payment request που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δούμε τότε κατά πόσο έχει αλλάξει το σύστημα. Ελπίζουμε βέβαια ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα πολλά προγράμματα όπου ακόμη έχουμε προβλήματα που πρέπει να διευκρινίσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αυτά θα αξιολογηθούν και θα αναπτυχθούν. Αυτή είναι λίγο πολύ απάντησή μου, αλλά επιτρέψτε μου ακόμη. Ασφαλώς θα σας δώσω αντίγραφο της ομιλίας μου, αλλά θα σας αποστείλουμε στο τέλος του μηνός και σχέδιο δράσεως θα το αποστείλουμε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα το διαβάσουμε και σε εσά για να δείτε ποια μέτρα λαμβάνει η κυβέρνησή μας για όλα αυτά τα θέματα έτσι ώστε να απλοποιήσουμε και να αλλάξουμε και την αντίληψη του συστήματός μας και να δείξουμε πώς θα βελτιώσουμε αλλά επίσης πώς θα τηρήσουμε τις προθεσμίες για κάθε μέτρο που θα εφαρμοστεί στο σύστημα. Θα σας τα διαβάσω λοιπόν έτσι ώστε να είμαστε και βέβαιοι και διαφανείς ότι όλα αυτά θα γίνουν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ Υπουργέ. Εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαι εγώ με τη Ρουμανία. Ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, ε, κάθε κυβέρνηση που ανέβαινε έπεφτε και ξανάβγαινε, μας ε, διαβεβαίωνε ότι θα άλλαζαν τα πράγματα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, αλλά θα ήταν ίσως καλό να κάνετε κάποια βήματα στα οποία έχετε δεσμευθεί ε, λέτε ότι τώρα εννοείται σοβαρά την καταπολέμηση της απάτης και της σύγκρουση συμφερόντων. Πόσους έχετε ε, μέχρι τώρα τιμωρήσει, πόσες κυρώσεις έχουν επιβληθεί, σε πόσα πρόσωπα από τότε που αναλάβατε. Γιατί γίνεται μεγάλη κριτική από τις εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά από μια τριετία παραγράφεται η απάτη και μάλιστα ε, δεν ε, διώκονται και ψηλές προσωπικότητες. Πότε σκοπεύετε στη Ρουμανία το χρόνο παραγραφής να τον διπλασιάσετε ή να πάει σε πενταετία ή σε εξαετία. Και το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο ε, σε ανώτατο επίπεδο έχει πρόβλημα και προσωπικού και χώρων. Αυτό πότε θα το αλλάξετε, πότε θα μεταρρυθμίσει το δικαστήριο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλε. Θα μπορούσατε ίσω να απαντήσετε αμέσω, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Θα ξεκινήσω από την τελευταία σας αναφορά, δηλαδή την έλλειψη προσωπικού. Και όσον αφορά τον αριθμό τους, αλλά και όσον αφορά την κατάρτιση που έχουν. Ακριβώς ε, σήμερα ε, έχω δημοσιοποιήσει ένα έγγραφο το οποίο αφορά το σχέδιο δράσης μας για την ε, ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας κυρίως των μονάδων που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή αναλύουμε σε κάθε επίπεδο, δηλαδή και στους ενδιάμεσους οργανισμούς και στους οργανισμούς διαχείρισης την κατάσταση για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει επάρκεια αριθμητική των ομάδων και αν η κατάρτιση των ασχολούμενων είναι αντίστοιχη με το ε, πεδίο με το οποίο ασχολούνται. Ε, διοργανώνουμε επαγγελματικές καταρτήσεις για το προσωπικό που εργάζεται Στι σε αυτές τις μονάδες, αλλά θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στις ειδικές αποστολές του προσωπικού, ας πούμε δημόσιες προσφορές, προμήθειες ε, και κάποια άλλα ευαίσθητα ε, θέματα. Θα στείλουμε ε, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με περιγραφή της κατάστασης αναμονάδα. Να δούμε ποιοι είναι οι εμπειρογνώμονες ε, για τις ε, δημόσιες προμήθειες, ποιοι είναι οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι είναι πάντα έτοιμοι έτσι ώστε να μελετήσουν τις καταστάσεις και τα ζητήματα που αφορούν τις προμήθειες, τις, την ε, ε, ε, και γενικώ όλοι αυτοί οι οποίοι μπορούν να είναι ανα πάσα στιγμή στη διάθεσή μας. Το πρόβλημα είναι ότι οι πραγματογνώμονες λόγω των χαμηλών μισθών που παίρνουν στο δημόσιο στρέφονται προς τον ιδιωτικό τομέα. Ε, θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τους μισθούς τους έτσι ώστε να τους κρατήσουμε στο δημόσιο ε, και θα ενισχύσουμε επίσης την επαγγελματική τους κατάρτιση. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στο δημόσιο. Όσον αφορά τις χειρώσεις... Μπορώ να πω το εξής. Όταν διαπιστώνουμε περίπτωση διαφθοράς, ο, ρόλος μας είναι να διαβιβάζουμε το ε, πρόβλημα αυτό, την υπόθεση αυτή στις ε, αρμόδιες αρχές. Έχουμε ε, μια ειδική αρχή για την καταπολέμηση της απάτης και εκείνοι κάνουν τις απαραίτητες έρευνες έτσι ώστε να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Εάν εμείς έχουμε κάποιες υποψίες όσον αφορά μονοεμένο άτομο ή ε, κατάσταση, τότε ε, ο εν λόγω υπάλληλος θα τεθεί σε διαθεσιμότητα θα σταματήσει λοιπόν τη δραστηριότητά του, ε, αν πρόκειται για μεμονωμένο άτομο και αν πρόκειται για ε, πρόγραμμα, ε, τότε δεν θα συμπεριληφθεί τα προγράμματα τα οποία θα αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι θα αποσαφινιστούν πολύ περισσότερο οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τώρα την περίοδο παραγραφής των αδικημάτων πρέπει να σας ομολογήσω ότι πρέπει να στραφώ προς τους αρμοδίους συναδέλφους και αργότερα θα σας αποστείλω σαφή απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τώρα τέσσερις ακόμα μιλητές και για να προλάβουμε θα πρότεινα να ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις. Έχετε ερώτηση επ' αυτού αμέσως τώρα κυρία Κρέσλε μετά ομαδοποίηση. Ναι, λέγει ο Υπουργός ότι έχουν ε, τεθεί σε διαθεσιμότητα κάποια αριθμό ρωτάω. Μπορείτε να μου δώσετε κανένα συγκεκριμένο αριθμό. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της δικιάς μου θητείας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 12, ε, θέσαμε σε διαθεσιμότητα μονάχα ένα άτομο. Και ε, αφορούσε ε, έναν ενδιάμεσο οργανισμό ε, που ισχολείται με ένα τμήμα του προγράμματος ανταγωνιστικότητας. Θέσαμε σε διαθεσιμότητα ε, το συγκεκριμένο άτομο που ήταν επικεφαλής, αλλά αποσύραμε και ολόκληρη την μονάδα η οποία ασχολείται με το ζήτημα αυτό, μέχρι ότου να κάνουμε τις απαραίτητες έρευνες. Ε, κοινοποιήσαμε την κατάσταση στο, στην Κομισιόν, την ειδοποιήσαμε δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι οποίοι εργάζονται στον ενδιάμεσο ε, φορέα ε, για την ώρα έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Τώρα θα ήθελα τέσσερις συνάδελφοι να μιλήσουν ο ένας μετά τον άλλον έτσι ώστε να έχουμε μια κοινή απάντηση εκ των υστέρων. Ο Ντι ε, Μούλντερ κλπ. Ε, ξεκινάμε με τον Ζωάν Πιέρο Ντι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την ε, παρουσία σας. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την πρωτοβουλία που ανέλαβε γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον συνάμα να έχουμε τέτοιες ανταλλαγές απόψεων σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω εγώ και το τονίζω αυτό, αναμένουμε πρόταση της κυβέρνησής σας ε, για τον ορισμό του ε, Ρουμάνου εκπροσώπου στο ελεγκτικό συνέδριο. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Έχει η κυβέρνησή σας πάρει θέση από αυτού. Ναι, να απαντήσετε μετά σε όλες τις ερωτήσεις. Γιάννη Μιλντερ. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου είναι μάλλον απλή. Έχουμε τις εκθέσεις του Ελληνικού Συνεδρίου, έχουμε και το, ε, ε τις εκθέσεις ε, του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συζητήθηκαν ε, στην χώρα σας. Ποια είναι η σχέση του δικού σας ελεγκτικού συνεδρίου σε όλη αυτή τη διαδικασία και ποια είναι η εκτίμηση του δικού σας ελεγκτικού συνεδρίου. Σένεγκαρντ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε ε, Υπουργέ και βεβαίως σας εύχομαι τα καλύτερα για τις ε, διαδικασίες και τις προσπάθειες που έχετε ξεκινήσει. Το 12 ξεκίνησε μια σειρά πρωτοβουλειών. Γιατί ε, ξεκίνησαν το 12 οι πρωτοβουλίες αυτές, ε, γιατί πολλά από τα προβλήματα είχαν ταυτοποιηθεί ήδη από πολλά χρόνια. Γιατί περιμένατε μέχρι το 12 έτσι ώστε να πάρετε αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμίλια, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ αναφερθήκατε σε μείζονος σημασίας μεταρρυθμίσεις στη Ρουμανία. Αλλά ένα από τα διαφορετικά προβλήματα στην Ρουμανία αφορά νέους ανθρώπους, ανθρώπους της δικιάς μου ηλικίας. Το πλαίσιο αλλάζει βέβαια, αλλά ε, τα πράγματα παραμένουν ίδια. Ε, διανύσαμε μία περίοδο σημαντικών πολιτικών αναταραχών και αυτό ε, δημιούργησε μεγάλη αγωνία και στρες στους νέους ανθρώπους. Όλη αυτή η διαρκής αλλαγή του πλαισίου, μάλλον αυτές οι διαρκείς αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν μια αγωνία στους νέους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν μετά από κάθε εκλογή να έχουμε ε, ε, αλλαγές ε, στα πάντα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια θεσμική ασφάλεια και παρακαλώ μην προδώσετε τους νέους που έχουν πιστέψει ε, σε αυτήν την ασφάλεια. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω απαντώντας την τελευταία ερώτηση. Ε, σας ευχαριστώ πάντως όλους για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση Μάλλον να σας το θέσω διαφορετικά. Λέτε ότι ε, κάθε κυβέρνηση τα αλλάζει όλα στη δομή του κράτους. Όχι. Ε, κάνουμε αλλαγές εκεί που αυτές ε, χρειάζονται. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε δομές οι οποίες δεν είναι σωστές και επίσης όσον αφορά τις οικονομικές δομές θα πρέπει να συζητήσουμε πριν πάρουμε τελικές αποφάσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις νοσιακές αρχές. Αλλάζουμε αυτό αυτά που ε, πρέπει να αλλάξουν. Είναι γεγονός ότι πρέπει να βελτιώσουμε το καταστατικό των, ε, ε, των υπαλλήλων, των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινοτικά κονδύλια. Αφού θα έχουν διοριστεί με διαφάνεια και σωστό τρόπο, θα πρέπει να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί μακριά από το πολιτικό φάσμα και τις πολιτικές ε, δραστηριότητες. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι αποτελούν εθνικό στόχο του οποίου θα πρέπει να υπεραμεινθούν όλες οι πολιτικές ε, δυνάμεις ε, και είμαι βέβαιος ότι τελικά αυτό θα συμβεί γιατί είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος με ρωτάτε γιατί πήραμε τα μέτρα το 2012 και όχι πιο πριν. Είναι γεγονός ότι η περίοδος αναφοράς είναι 2009-2011. Δυστυχώς είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα στην περίοδο αυτή 2009-2011 ε, και η Κομισιόν σημείωσε τις ε, ανομαλίες ε, για όλη την περίοδο 9 με 11 αλλά λόγω της ε, ε, κατάστασης δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. Όμως από το 2012 και μετά η Ρουμανία ε, δέχτηκε να πάρει συγκεκριμένα μέτρα και τώρα καταβάλει πλέον όλες τις προσπάθειες έτσι ώστε να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς επίσης και τα κράτη-μέλη ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι αλλάζουν τα πράγματα στη Ρουμανία, ότι θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση. Θέλουμε το 2013 να αποτελούμε πρότυπο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον όσον αφορά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να το κάνουμε και έχουμε τη βούληση να το κάνουμε. Για να απαντήσω τώρα στην άλλη ερώτηση, η οποία αφορά τη σύγκριση ανάμεσα στην έκθεση του ελεγκτικού ε, συνεδρίου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, το με την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου της Ρουμανίας. Αν κατάλαβα καλά αυτό με ρωτήσατε. Και εγώ έχω δουλέψει στο ελεγκτικό συνέδριο της χώρας μου. Μπορώ να σας πω ότι έχει γίνει αυτή η σύγκριση και είναι πάρα πολύ χρήσιμη μάλιστα, γιατί όλες οι συστάσεις ε, του οικονομικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου λαμβάνονται υπόψη για κάθε σύσταση το Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο ε, ε, ε, κάνει αντιστοίχως κάποιες συστάσεις και παρακολουθεί την υλοποίηση των συστάσεων σε όλη την πορεία της διοικητικής αλυσίδας. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει στη διάθεσή του όλες τις συστάσεις που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ε, και από τους εξωτερικούς ελεγκτικούς ε, οργανισμούς. Ε, και το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ρουμανίας κάνει τις τελικές διακριβώσεις. και εγώ ο ίδιος έχω ζητήσει να γίνονται τέτοιες διακριβώσεις σε, όλα τα στάδια, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε ε, το σωστό έλεγχο των συστάσεων, διότι έχουμε βρει ε, συστάσεις οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί ε, τελικά. Αυτό που θέλουμε, το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να υλοποιηθούν όλες οι συστάσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί. Η τελευταία ερώτηση τώρα, αυτή η οποία αφορά ε, τον ε, ορισμό του ε, Ρουμάνου εκπροσώπου στο ελεγκτικό συνέδριο. Πρέπει να σας πω ότι πολύ σύντομα θα προτείνουμε ένα όνομα. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, ξέρουμε ότι πρέπει να ορίσουμε κάποιον άλλον. Γνωρίζουμε ότι οι διακριβώσεις παίρνουν και οι επαληθεύσεις παίρνουν χρόνο. Πάντως, ε, πάρα πολύ σύντομα η Ρουμανία θα προχωρήσει ε, στον ε, διορισμό. Και είμαι σίγουρος ότι το άτομο το οποίο θα προτείνουμε θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και προϋποθέσεις για την κάλυψη της αυτής. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Είναι και χαρά και τιμή που σας είχαμε σήμερα μαζί μας ε, βλέπετε ότι παρά τις επίμονες ερωτήσεις, δύσκολες ερωτήσεις, έχουμε και επικοδομητική ε, προσέγγιση. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ, ευχαριστούμε που απαντήσατε στα ερωτήματά μας και βεβαίως ελπίζουμε σε περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων. Ε, ο κύριος Θεοντοροβίτσι, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Είμαι ανοιχτός για οποιασδήποτε, ε, προσθε... Ε, οποιασδήποτε ε, ερωτήσεις. Μπορώ να απαντήσω και αργότερα στις ερωτήσεις τις οποίες θα μου θέσετε ενδεχομένως. Ευχαριστώ πολύ. Ich unterbreche die Sitzung Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα. 4 προσοχή, όχι 3.